Πες τα we have five minutes. Πέντε λεπτά μας έχουν απομείνει. Στις μία ακριβώ πρέπει να ολοκληρώσουμε. Περνάμε στο σημείο 12, το τελευταίο της πρωινής μας συνεδρίασης. Σύναψη συμφωνίας για την ε, αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ε, Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας. Συντάξαμε έκθεση με τη μορφή επιστολής που θα ψηφίσουμε το απόγευμα κατά το τέλος συνεδρίασης. Ε, μάλιστα, με την γραπτή διαδικασία στις 10 Ιανουαρίου οι συντονιστές έδωσαν το πράσινο φως και σας στείλαμε ε, την επιστολή λίγο αργότερα. Συστήνουμε στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συστήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει την έγκρισή του για τη διαδικασία περί αποχώρησης με βάση τα άρθρα 127, 129 και 156. Στις 23 ε, ε, Ιανουαρίου η ΑΦΚΟ θα ψηφίσει για την συγκατάθεση και στις 29 Ιανουαρίου στη Μήνη Ολομέλεια των Βρυξελών ενημερώθηκα ότι θα κατατεθεί στην παράγραφο 1 προφορική τροπολογία της ομάδας των φιλελευθέρων του Ρινιού ε, για να προσθεθεί και το λυπούμαστε, we regret. Σύμφωνα με την πρόταση της ομάδας Ρινιού. Γιατί φυσικά με βαθύτατη λύπη παρακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις, οπότε το ε, εκφράζουμε τη λύπη μας, ε, είναι αποδεκτή η τροπολογία. Η κυρία Φομβίζε. Γνωρίζω ότι έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τις συζητήσεις που είχαμε στην ομάδα και γιατί είναι πολύ δύσκολο για μας τους ευρωβουλευτές του Ηνωμένου Βασιλείου να εγκρίνουμε την επιστολή παρά την προσθήκη του ε, We regret ή με, με έκφραση θλίψης ή εκφράζουμε τη θλίψη μας. Η Βρετανική Αντιπροσωπεία και φαντάζομαι και άλλοι πιστεύουμε πως και άλλοι ότι αυτή η συμφωνία περί αποχώρησης δεν είναι σωστή και δεν δίνει τα απαραίτητα για, για το συμβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών και επίσης ε, ε αφήνει ανοιχτή την ε, πιθανότητα ε, για ένα Brexit χωρίς, συμφωνία προς τα τέλη του μήνα και με το τέλος της προθεσμίας μάλλον και γι' αυτό δεν μπορούμε να δώσουμε τη συμφωνία μας στην επιστολή και ελπίζω να μην περάσει την ψηφοφορία. Βέβαια, οι συγκεκριμένες τροπολογίες για συγκεκριμένες συστάσεις που αφορούν τις ε, ε, εξωτερικές σχέσεις είναι πολύ σημαντικές και πολύ εύστοχες προσθήκες, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορώ να ψηφίσω οτιδήποτε αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, για την οποία όχι μόνο λυπούμε βαθύτατα, αλλά θεωρώ ότι είναι και ολέθρια. Είναι η Ναγγέλ. Ευχαριστώ. Εστενίζουμε πλήρως τα λεγόμενα της προλήσης και η αντιπροσωπή των εργατικών του Ηνωμένου Βασιλείου. συμφωνούμε ε, ότι ήταν προβληματική η συμφωνία περί αποχώρησης και πόρο απέχει από τις συζητήσεις που είχαμε στη Λιόν. Θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις παρόλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, μια και είστε ο εισηγητής, συντάκτης αυτής της επιστολής. Ποιο θα είναι το μελλοντικό σενάριο, γιατί μιλάτε για την κοινή ε, πολιτική ασφάλειας και άμυνας και την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα αυτά στο μέλλον. Θα έχουμε κάτι συγκεκριμένο για την πιθανή συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε αυτές τις δύο πολιτικές. Βέβαια, σε αυτή τη φάση δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως ε, αυτό το ενδεχόμενο. Πάντως, η Βρετανική Αντιπροσωπεία ε, πολύ πιθανόν να μην υπερψηφίσει την επιστολή για την έγκριση της Συμφωνίας περί αποχώρησης. Ευχαριστώ. Μάρκ, ευχαριστώ. Και θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με την προφορική τροπολογία του Ρινιού να προσθεθεί, εκφράζει την θλίψη του. Θα συμφωνούσα με τη δική σας πρόταση, εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του, γιατί το Brexit είναι κακό και για την Ευρώπη και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Και παρόλο που η επιστολή είναι εξαιρετική και τονίζει την ανάγκη συνεχούς ε, στενής συνεργασίας για θέματα ασφάλειας και άμυνας, ε, για τα πρακτικά θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με την κυρία Φομβίζη ότι η ίδια συμφωνία περί παραχώρηση για την οποία θα πρέπει να δώσουμε τη συγκατάθεσή μα, είναι πολύ κακή και δεν προστατεύει δεόντω του πολίτε των 27 χωρών και τα δικαιώματά του για τη Βρετανία μετά τον Brexit και για τη Βόρεια Ιρλανδία προβλέπει περίπλοκες ε, διατάξεις, ε, ίσως και δύσκολες εφαρμογής για να αποφευθεί το σκληρό σύνορο μεταξύ Βόρειο Ιρλανδία και Ιρλανδία και απειλεί τη μελλοντική ασφάλεια και ειρήνη εκεί. Και επίση, παρά την ε, πιθανότητα ε, συνθηκών ισότιμου ανταγωνισμού μεταξύ Βρετανία και Ηνωμένου Βασιλείου, στην πολιτική διακήρυξη, που δεν είναι δεσμευτική για τα μέρη, ε, αναφέρεται αυτό. Οπότε υπάρχει άμεση απειλή για τα εργασιακά τα δικαιώματα, τι προδιαγραφέ και τα πρότυπα για τι κρατικέ ενισχύσει και το περιβάλλον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και υπάρχει διαφορά μεταξύ των πρότυπων αυτών και των πρότυπων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπω έτσι λοιπόν ε, δημιουργώντα μια οικονομία στο Ηνωμένο Βασίλειο τύπου Τραμπ, δημιουργηθεί στρέβλωση ανταγωνισμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ αρνητική λοιπόν η συμφωνία για τη Βόρεια Ιρλανδία, την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ και εδώ δυστυχώ διακόπτεται η διερμηνία. Το απόγευμα θα συνεχιστεί η συνεδρίαση και θα γίνει και η ψηφοφορία. The η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει το, την εντολή για την επόμενη φάση το Φεβρουάριο. Το Συμβούλιο θα εγκρίνει αυτή την εντολή στις 25 Φεβρουαρίου και εμείς στο μεταξύ θα εγκρίνουμε το ψήφισμα στην συνεδρίαση του Στρασβούργου είτε 12 είτε 13 Φεβρουαρίου. και εκεί θα αναφέρουμε τις κατευθυντήριες γραμμές μας. Εδώ δυστυχώς θα πρέπει να σταματήσει η διερμηνία. Καλώς σας μεσημέρι. transition period and I believe that the Commission President set the tone at her speech at the LSE. If we only have a limited time frame,